επίσημη στην ιστοσελίδα του διαδικτύου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το ημερήσια διάταξη και τώρα περάτε των εργασιών μας για απόψε. Καλώς βράδυ.